Γεια σας. Καλό από μεσημερό. Μόλον ότι είμαστε όλοι γάριθμοι. Ήδη πέρασε ένα τέταρτο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τις εργασίες της Επιτροπής. Ας περάσουμε το πρώτο σημείο της ημερησίας που είναι η έγκριση της ημερησία διατάξεως ε, που αναμφίβολα έχουν δει οι συνάδελφοι. Μοναδικό αίτημα τροποποίηση που έχει υποβληθεί είναι αυτό της αντιστροφής των σημείων 15 και 16. Ε, θα τα εξετάσουμε από το πρωί. Το αίτημα πρόκειται από τον συνάδελφο Βαλέσα για λόγους ηλεμένων υποχρεώσεων ζητάει να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα του πριν από το θέμα του συναδέλφου Σαλαβράκου ο οποίος με ενημέρωσαν ότι δέχθηκε αυτή την αλλαγή. Άρα λοιπόν θα προταχθεί το θέμα του κύριου Βαλέσσα σε σχέση με το θέμα του κύριου Σαλαβράκου. Έχουμε τους αναφερόμενους για τις 446, 684 ε, του 2012, στο σημείο 10 είναι γραμμένες, στο σημείο 20 είναι μια άλλη αναφορά για το εγκαταστάσεις του Βουκουρέστη και μια άλλη που αφορά στο σημείο 21 δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις Θεωρούμε ότι εγκρίνεται η μισή δεν υπάρχουν στάσεις. Στο σημείο 2 έχουμε την έγκριση των πρακτικών των δύο συνεδριάσεων της 25-26 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν στάσεις, ε, όχι. Άρα εγκρίνονται και τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Μπορούμε λοιπόν με τρόπο αυτό να περάσουμε στο πρώτο σημείο της μεσαίας διάταξης. Πρόκειται για την αναφορά 446-2007 που έχει υποληθεί από τον Βρετανό υπήκο σχετικά με το δικαίωμα της ψήφου στις εκλογές για την Εθνικό Κοινοβούλιο της Αγγλίας για τους εγκαριστημένους στο εξωτερικό. Ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν, αλλά είναι παρούσα η κυρία Σαρλότ Όλιβερ. Έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Thank you very much. Uh, I'm representing... Ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπο των Χαρισίλ εδώ σήμερα. Ήθελε πολύ να παρευρίσκεται εδώ, αλλά είναι 93 ετών και Αγωνίστε για αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Το 2007 έκανε την αναφορά και μετά είχε προτεραιότητα η αίτησή του στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 2013 αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι Βρετανοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό για πάνω από 15 έτη δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να ψηφίζουν σε εθνικές κοινοβουλευτικέ εκλογές. Ο Χαρή θεωρεί ότι αυτό αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος του υπό το άρθρο 3.1 της συνθήκης. Εξετάστηκε προσεκτικά το θέμα. Πέντε χρόνια προηγουμένως υπήρχε η υπόθεση Ντόιλ επί του ίδιου θέματος. Παρότι το Μάιο πέρυσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι δεν υπήρχε παραβίαση, διότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μόνο τους δικούς του εκλογικού κανόνες. Εφόσον αυτό γίνεται για θεμητό σκοπό για να οριστεί δηλαδή κατά πόσο υπάρχει η σχέση του εν λόγω ατόμου με την χώρα πρόέλευση, Λένε ότι το μέτρο αυτό είναι αναλογικό, Συνεπώ δεν αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων ενό ατόμου. Στη συνέχεια, ο Χαρή μαζί με εμένα και μια αντιπροσωπή άλλων Βρετανών πολιτών που ζουν σε διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε στην Κομισιόν τον Σεπτέμβριο και μίλησε απευθεία με τη Vivian Ρέντινγκ, που όπω γνωρίζετε πέρυσι ε, προέβησε πολύ θετικά σχόλια που υποστήριζαν την υπόθεση του Χάρι Σέντλερ. Ε, ανέφερε ειδικότερα ότι θεωρεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο αρνούμενο το δικαίωμα ψήφου στις κοινοβουλευτικές εκλογές ε, πολίτες του που διαμένουν στο εξωτερικό για πάνω από 15 χρόνια ουσιαστικά είναι σαν να τιμωρεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας αυτός ο κανόνα ισχύει και για μένα. Εγώ είμαι Βρετανίδα ε, υπήκος, ε, δικηγόρος και διαμένω στην Ιταλία. Και όπου εργάζομαι ως αβοκάτο με πλήρη δικαιώματα εργασία εκεί, αλλά διατηρώ τα, σε με το Ρωμανό Βασίλειο. Το 90% των πελατών στην Ιταλία είναι Βρετανοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό ή που έχουν ιδιοκτησία στο εξωτερικό. Από το 2016 λοιπόν αυτός ο κανόνα θα καλύπτει και εμένα και παρότι εγώ εκπροσωπώ βρετανου πολίτε καθημερινά πρέπει να του εξηγήσω τις ε, διαφορές μεταξύ Ιταλικού και Βρετανικού δικαίου και τελικά θα χρειαστεί να απολέσω και εγώ το δικαίωμα ψήφου μου. Πιστεύω 1,7 ε, εκατομμύριο Βρετανοί πολίτες διαμένουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη και αυτό θα ισχύει για όλους αυτούς. Μετά από τη συνάντησή μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπω αναγραφεί σχετική έκθεση, για να ορίσει αυτόν τον κανόνα ως ε, κανόνα που εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση. Ε, ο Χαρή σα ευχαριστεί για την πρόσκληση εδώ. Επτά χρόνια αφού υπέβαλε την αναφορά και η αναφορά κανονικά δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο για να φτάσει στην Επιτροπή αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι η περσινή απόφαση και τα σχόλια της Βεν Ρέντινγκ επανέφεραν στο προσκήνιο το θέμα αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για Βρετανούς πολίτες ε, που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο δημοψηφίσματος από το 2015. Τώρα περνάει από τη Βουλή. Δημοψήφισμα για το κατά πόσο το Ηνωμένο πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Άνθρωποι όπως εγώ και ο Χαρίς Σίντλερ σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουν το δικαίωμα ψήφου σε ένα τέτοιο δημοψήφισμα παρότι εμείς έχουμε ε, από πρώτο χέρι εμπειρία για το πώς αυτή η ελευθερία που παρέχεται στους Ευρωπαίους πολίτες λειτουργεί στην πραγματικότητα όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και ε, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε την άποψή μας για το κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη ή όχι. Αυτό επηρεάζει και άλλες χώρες πέντε κράτη-μέλη, Γερμανία, Ιρλανδία, Δανία, Κύπρος και Μάλτα. Και, σε κα... και αυτές οι χώρες σε κάποιο βαθμό περιορίζουν τα δικαιώματα ψήφου για τους ε, ε τους που κατοικούν εκτός αυτών των χωρών. Δηλαδή αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου για αυτά τα άτομα μετά από κάποιο ε, χρόνο διαμονή στο εξωτερικό. Ο Χαρισίντλερ ε, κατοικεί στην Ιταλία εδώ και σχεδόν 13 χρόνια. 30 χρόνια, συγγνώμη, και έτσι του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα ψήφου. Δεν έχει πλέον το δικαίωμα ψήφου λοιπόν. Αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση, αποτελεί αφαίρεση των δικαιωμάτων ψήφου, διότι όχι μόνο δεν έχει το δικαίωμα ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το έχει ούτε στην Ιταλία. Όπω προτείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει την επιλογή να γίνει Ιταλό υπηκό, εάν επιθυμεί να ψηφίζει στη χώρα όπου διαμένει. Ήταν πολύ δυσάρεστο να ακούει κανεί κάτι τέτοιο. Η υπηκότητα είναι ο πρώτο σύνδεσμο που έχουμε με τη χώρα μα, με την κοινωνία, με την πολιτική τη και πρέπει να αποφασίζουμε εμεί οι ίδιοι κατά πόσο θα δίνεται αυτή η σύνδεση. Θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα ψήφου στη χώρα προέλευσή μα, διότι διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να επιστρέψουμε σε αυτή τη χώρα και να ζήσουμε εκεί. Έχουμε λοιπόν αυτή την ομάδα Βρετανών πολιτών και άλλων πολιτών που διαμένουν στην Ευρώπη και καλούμε να εξεταστεί το θέμα πριν από τις επόμενες ε, Βρετανικές εκλογές το 2015, πριν από ένα πιθανό δημοψήφισμα στο οποίο θα μας απαγορεύεται η ψήφος. Ζητάμε από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες της αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξαναδεί αυτό το θέμα, να υποβληθεί ένα ψήφισμα για να μπορέσουμε να δούμε εμείς ως πολίτες τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Ζητήσαμε να παραπαινθεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παρότι σπανίζουν οι υποθέσεις αυτής της, αυτού του είδους να παραπέμπονται από την Κομισιόν στο Δικαστήριο ζητάμε σε αυτή την περίπτωση όπου είναι σαφής ε, ξεκάθαρη η διακριτική μεταχείριση και τιμώρηση ανθρώπων που ασκούν το δικαίωμα ε, ελεύθερη κυκλοφορία. Ζητούμε λοιπόν αυτό το θέμα να εξεταστεί κατεπήγον. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Όντω, Όπω είπε η ε, κυρία που εκπροσωπεί τον αναφερόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γνώση αυτού του φαινομένου. Σήμερα κανένα κράτος μέλος δεν χορηγεί ε, το δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές σε επικόους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην επικράτειά τους. Ε, τους έχει αφαιρεθεί λοιπόν το δικαίωμα και δεν μπορούν να ψηφίζουν πουθενά σε βουλευτικές εκλογές, ούτε στη χώρα τους ούτε σε εκείνη την οποία διαμένουν. Αυτό βέβαια δεν συνάδει με το γεγονός ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή. Από την άλλη όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διοργάνωση εθνικών βουλευτικών εκλογών είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Οποιοδήποτε μέτρο και να λάβουμε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονός αυτό. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους για το ζήτημα αυτό και τελικά το 2013 στην αντίστοιχη έκθεση για την Ιθαγένεια ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προτείνει επικοδομητικού τρόπου έτσι ώστε πολίτε τη Ένωση που διαμείνουν σε άλλη χώρα από την πατρίδα του να διατηρούν το δικαίωμα ψήφου στι βουλευτικέ εκλογέ στην χώρα προέλευση. Τα νέα λοιπόν που μπορώ εδώ τώρα σήμερα να σας ανακοινώσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σύντομα θα καταθέσει πρόταση και θα προτείνει αυτά τα επικοδομητικά μέτρα και στις αρχές του 2014 θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα στους ερχόμενους μήνες και εβδομάδες ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να λάβει το λόγο περί του θέματος. Ε, από ό,τι φαίνεται όχι. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή η αναφορά ε, αναφέρεται σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ήδη γνωστό από τους συναδέλφους όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μόνο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης διότι το θέμα αφορά εθνικό ζήτημα και την, εθνική, και την νομοθεσία περί συμμετοχής εθνικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, μετά την πρωτοβουλία την οποία πρόθεσε η Επίτροπος Ρέντινγκ, το θέμα ε, βρίσκεται στην, ε, υπό τη, στην υπαρακολούθηση, θα λέγαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι προφανές ότι υπάρχει παραβίαση ε, δικαιώματος των πολιτών προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν πάντα και οπουδήποτε το ενεργητικό και υποθετικό δικαίωμα στις εκλογές και αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Ως εκ τούτου μπορεί να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να προχωρήσουμε με τις εργασίες που εδώ και χρόνια ο κύριος Σίντλερ έχει ξεκινήσει από πλευράς του προσπαθώντας με ένα περαιτέρω σημείωμα να ζητήσουμε από την Επίτροπο Ρέντινγκ και από την Κομισιόν να επιταχύνουν το βήμα τους ε, προς την κατεύθυνση που, έχει ήδη που έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν δεν υπάρχουν αντίθετες απόψεις, ε, ούτως θα πράξουμε. Ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Όλιβερ που μας παρουσίασε την αναφορά του κυρίου Σίντλερ. Παραμένει ανοιχτή. Θα γράψουμε στην Επιτροπό Ρέντινγκ προκειμένου να ζητήσουμε στήριξη του δικαιώματος της ψήφου όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Περνάμε στο επόμενο ζήτημα της μισής διάταξης. Πρόκειται για την αναφορά που αναφέρεται στο σημείο 6, αναφορά 1138-2012 από πλευρά ενό Έλληνα υπηκόου, εξ των ταξιδιωτικών λεωφορείων κεντρική και βόρειας Ελλάδας αναφορικά με την απελευθέρωση των οδικών επιβατικών μεταφορών. Δεν είναι παρόν ε, ο αναφερόμενος. Ε, ας ακούσουμε την γνώμη της ε, Κομισιόν και δίνω το λόγο στον κύριο Μικού. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη. Ε, είδατε την απάντηση της Κομισιόν 2013, ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε ήδη αναλάβει διαβήματα για να απελευθερώσει τις οδικές υπηρετικές μεταφορές στην Ελλάδα και ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο ότι σε ό,τι φορά τους χειρισμούς περί φορολογικών απαλλαγών και εκτιμάτων, η Κομισιόν εξετάζει ήδη το ζήτημα. Από τότε, ειδικά την 1η Οκτωβρίου 2013, η Ελλάδα υιοθέτησε ένα νόμο πλαίσιο για την απελευθέρωση των οδικών βιωτικών μεταφορών στη χώρα και μερικές εβδομάδες αργότερα ε, ολοκληρώθηκαν οι ενέργειές μας αναφορικά με την συγκεκριμένη αναφορά ε, ε, διότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν δεν βρήκαν καμία παραβίαση των κανόνων και της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ε, κάποιος ζητάει το λόγο. Ουδής ε, θέλει να λάβει το λόγο. Κύριος Σαλαβράκος. Ε, εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι επειδή δεν υποστηρίζεται από πλευράς του ετούντος και επειδή βεβαίως ε, έχει απελευθερωθεί το επάγγελμα των οδικών επιβατικών μεταφορών θα κρίνω επαρκής τις, ε, ε, τις σημειώσεις της Κομισιόν. Ο συνάδελφος Σαλαβράκος ζητάει να κλείσει η αναφορά. Έτσι δεν είναι. Επίσης. Δεν υπάρχουν στάσεις από πλευρά συναδέλφων. Ε, από το ιστορικό της αναφοράς προκύπτει ότι η Κομισιόν ε, άνοιξε μία έρευνα σχετικά με την αναφορά του Βασίλειου Αντανόπουλου και η εξέλιξη της έρευνας ε, έφτασε μέχρι την σήμερα και η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα απελευθέρωσης τα οποία ικανοποιούν τις ε, επιθυμίες του Έλληνα αναφερόμενου και όπως είπε ο κ. Σαλαβράκος ολοκληρώνεται εδώ η εξέταση αυτής της αναφοράς ελπίζοντας πως η κατάσταση με τα νέα αυτά μέτρα που έλεγε η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να επιληθεί. Ολοκληρώνεται λοιπόν η εξέταση αυτής της αναφοράς. Περνάμε στην ε, Αναφορά 712, 711 συγγνώμη το 2012 από μια Πολωνή ε, πίκο από του Δικηγόρου Γραφείου Καντσελάρια Πράουελ Βίγκεν σχετικά με την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του κανονισμού αριθμό 1071-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά του όρου που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματο του οδικού μεταφορέα και την κατάργηση τη οδηγία 96-26 του Συμβουλίου. Αναφέρον εκφράζει την άποψη ότι η πολωνική νομοθεσία δεν τηρεί, το πολωνικό δίκαιο δεν τηρεί την ε, σχετική νομοθεσία και δίνω το λόγο λοιπόν στον υπεύθυνο της Κομισιόν Σασίμσκα. Αδύνατο να προφέρω σωστά το όνομά σας από ό,τι φαντάζομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο από την αναφορά κατάλαβα ότι το νομικό γραφείο που εκπροσωπεί ο αναφερόμενος ε, δεν μιλάει για παραβίαση από την πολιτική κυβέρνηση αυτού του νόμου απλά δεν συμφωνεί με τη διατύπωση στο παράρτημα 4 λέει ότι δεν είναι σαφές όπως ε, λέει η απάντηση στην αναφορά, η διατύπωση στο παράρτημα 4 όπου αναφέρεται μια λίστα των πιο συχνών παραβιάσεων των κανόνων οδικών μεταφορών δεν είναι ακριβώς ίδια όπως στη βασική νομοθεσία στην οποία αναφέρεται. Όπως εξηγήθηκε, διευκρινίστηκε αυτή η περιγραφή των πιο συνήθων παραβιάσεων που προβλέπεται στο παράρτημα 4 του κανονισμού 1071 θα πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο του κανονισμού 561 για τις ώρες εργασίας και τις ώρες ανάπαυσης των οδηγών. Αυτός ο κανονισμός ουσιαστικά δεν αναφέρεται αυτός καθεαυτός στον κανονισμό 1071 που αποτελεί το αντικείμενο αυτής εδώ της αναφοράς. Ωστόσο στο άρθρο 6.1 του 1071 γίνεται αναφορά στου κοινωτικούς κανόνες στους τομείς μεταξύ άλλων των ορών οδήγηση και των ορών ανάπαυσης των οδηγών. Αυτό, ο κανονισμό, ο 561 ε, αναφέρει αυτούς τους κανόνες, περιλαμβάνει αυτούς τους κανόνες, ε, ο 561 του 2006 για τους οδηγούς. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο το 1αβ του 1071 έχει διατυπωθεί πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισμού 561. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος το λόγο. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Για το έτοιμο λοιπόν του αναφερόμενου ουσιαστικά ζητά ποια είναι η σωστή ερμηνεία τη νομοθεσία στην οποία αναφέρεται. Εγώ θεωρώ ότι δεδομένη τη απάντηση που μα έδωσε τώρα η πρόσωπο τη Κομισιόν, μπορούμε και να κλείσουμε την αναφορά αυτή. αποσταλώντα ε, στον αναφερόμενο και στου πολίτε που εκπροσωπεί αυτό ε, την σημερινή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας ε, δίνει μια κατεύθυνση για το πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε σωστά τα νομοθετικά κείμενα ε, που θεωρούνται σύμφωνα με την αναφορά όχι πολύ σαφή ώστε να λυθεί το πρόβλημα συγκεκριμένης ε, υλοποίησης που οφείλεται στο πρόβλημα ερμηνείας. Αν δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις να στείλουμε αυτή την ερμηνεία στον αναφερόμενο τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να κατανοήσει τους ε, κανόνες έτσι όπως το προτείνει η Κομισιόν. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Κλείνουμε λοιπόν ε, την ε, αναφορά. Παίρναμε τώρα στην αναφορά 8. 0021 του 2013 του κυρίου Τζον Σαβάτζ, Βρετανικής Ιταγένειας σχετικά με τις υπέρμετρες δαπάνες του Πάρκου Διαχείρισης ε, Αποβλήτων Άλλαρτων. Και στην αναφορά παρουσιάζει κάποιες ε, αιτίες. Ε, να ακούσουμε την Κομισιόν, διότι ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντίας Δελκαστήγιο. Στα αγγλικά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή έχει να κάνει με περιβαλλοντικά ζητήματα και ε, τις κρατικές ενισχύσεις στον ανταγωνισμό δηλαδή και τις δημόσιες συμβάσεις. Τρεις είναι οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις που ενέχονται εδώ. Εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και θα περιοριστώ στις περιβαλλοντικές ενδεχομένως πτυχές και αντίκτυπο αυτού του έργου. Στη συνέχεια άλλο συνάδελφος θα αναφερθεί στα υπόλοιπα. Πρώτον, ε, το έργο που περιγράφει αναφορά Ε, ε, έχει να κάνει με μια μονάδα αποτέφρωσης ε, και μηχανικού διαχωρισμού και παραγωγής θερμότητας. Είναι στο στάδιο ακόμα του σχεδιασμού του έργου και εξ όσων γνωρίζουμε από τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο αναφερόμενος δεν έχει δοθεί ακόμα η οικοδομική άδεια. Δεύτερο, ο αναφερόμενος αναφέρεται ε, στο θέμα της δυνατότητας αποτέφρωσης εκεί και της ιεραρχίας των ε, διαφόρων αιτημάτων. 49% ε, των αποβλήτων το 2011 στο Ηνωμένο Βασίλειο πηγαίναν σε ε, χωματερές. Το 39% ανακυκλώνεται και το 12% αποτεφρώνεται. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, 12 κράτη-μέλη ε, αποτεφρώνουν περισσότερο από το 12% αυτό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με πρώτη τη Δανία που αποτεφρώνει το 54% των στερεών αστικών αποβλήτων. Αυτό είναι σημαντικό για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια είναι η ιεραρχία στην ανακύκλωση, ε, η ανακύκλωση, η αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να είναι μια καλή επιλογή ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μη ανακυκλώσιμα απόβλητα για να μην καταλήξουν στις χωματερές σε χιτά. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, συνολικά δεν έχει ε, τις δυνατότητες που έχουν η Δανία και η Σουηδία ως προς την αποτέφρωση. Ε, για να συμπεράνω, αν προχωρήσει αυτό το έργο, μάλλον ε, θα υπόκειται στην οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν φτάσει στο στάδιο λειτουργίας υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές ρήπων. Άρα τα στοιχεία αυτά του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας θα ληφθούν υπόψη και ε, θα ε, καλυφθούν από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Σίλβα. Thank you very much, Chair. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο αναφερόμενος θέτει δύο βασικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ορθότητα Τη διαδικασία για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το πρώτο θέμα αφορά το ότι δεν έχουν παρασχεθεί επαρκείς πληροφορίες από την αρχή. Αυτό μπορεί να αποθάρρυνε κάποιους πιθανούς ε, αναδόχους να προσφέρουν καμιά προσφορά για το έργο. Η ειδοποίηση για τη σύμβαση αναφερόταν μόνο σε αστικά απόβλητα και όχι σε εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα που εντάχθηκαν στο Συμβόλαιο σε μεταγενέστερο στάδιο. Παρ' όλα αυτά εμείς ε, δεν θεωρούμε ότι τίθεται θέμα παραβίασης ή παρανομίας. Εάν κοιτάξετε τους κωδικούς στην ειδοποίηση σύμβασης για αυτή τη συγκεκριμένη σύμβαση γινόταν αναφορά στο πλαίσιο του λεξιλογίου κοινών προμηθειών ε, κάτι που αναφερόταν στα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα υπό τους κώδικες λοιπόν σε επειδή δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα θεωρούμε λοιπόν ότι όποιοι οικονομικοί φορείς ε, θα ενδιαφέρονταν να κάνουν προσφορά για αυτό το συμβόλαιο, για αυτή τη σύμβαση, δεν πρόκειται να αποθαρρυνθούν από το γεγονός αυτό. Δεύτερον, ο αναφερόμενος αναφέρεται επίσης στη μεγάλη διάρκεια 25 έτη της ε, σύμβαση. υπό την ισχύουσα οδηγία 2014-17 για τις δημόσιες προμήθειες δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια για τις συμβάσεις. Δεν βλέπουμε λοιπόν ούτε εδώ να υπάρχει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ήθελα επίσης να αναφερθώ στο γεγονός για να κλείσω ότι ο αναφερόμενος αμφισβητεί την επιλογή της τεχνικής λύσης και την αγορά ενός πολύ ακριβού αποτεφρωτή για τη συμβασία αυτήν. Οι κανόνες δημοσίων συμβασιών αφορούν τον τρόπο αγοράς και όχι το αντικείμενο αγοράς. Η συμβάλλουσα αρχή λοιπόν είναι αυτή που αποφασίζει τι θα αγοράσει. Βαλόμενη αρχή, συγγνώμη. Ζήτησε κάποιο το λόγο. Κύριο Γιάρ. Ναι. Μια συμπληρωματική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τα γνωρίζω από δική μου εμπειρία για το τι γίνεται με τη διάθεση των αποβλήτων και ε, ο εξοπλισμός και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν και ανάβουν τα αίματα και φωνάζουν οι πολίτες, ε, ε, λένε οι πολίτες ότι αυξάνεται το κόστος και κατηγορούνται οι εταιρείε ότι βγάζουν πολλά λεφτά. Τα γνωρίζω λοιπόν αυτά από ίδια πείρα. Και ε, ξέρω ότι ε, εκφράζονται επικρίσεις για το χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Πρέπει να γίνει μια διάκριση. είναι μόνο η συλλογή και η αποκομιδή. Αυτό μπορεί να είναι σύντομο διάστημα. Αλλά όταν κάποιος ε, θέλει να εγκαταστήσει ε, μονάδα αποτέφρωσης θα πρέπει να έχει ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να προκυρήσετε για μία πενταετία μόνο το έργο γιατί είναι βαριά υποδομή και μετά από πέντε χρόνια που θα το έχει κατασκευάσει ο άλλος ε, είναι ερήπιο επενδυτικό. Εσείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπετε να έχουν παραβιαστεί νόμοι που έχουν να κάνουν με την προκήρυξη του έργου. Περί αυτό πρόκειται. Το ξέρω ότι αυτός που αναλαμβάνει το έργο μπορεί να ορίσει τι θα κάνει ή και κάθε περιφέρεια, κάθε χώρα, πώς θα ανακυκλώνονται, ακόμα και σε ποια εταιρεία θα ανατεθεί το έργο, το αποφασίζουν οι αρμόδιοι φορείς. Αυτά είναι όλα εντάξει. Αλλά η αναφορά έχει να κάνει με το εξή. Κατά την άποψή σας έχουν παραβιαστεί οποιασδήποτε οδηγίες σχετικές με την προκήρυξη διαγωνισμών για δημόσιες προμήθειες. Αν μας πείτε όχι, μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Αν μας πείτε δεν το γνωρίζω, δεν έχω αρκετή ενημέρωση, θα πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή αναφορά. Για μένα αυτό είναι το αποφασιστικό και όχι ζητήματα τώρα τεχνικά ουσίας. Από ό,τι φαίνεται εσείς ε, πιστεύετε ότι έχουν γίνει όλα σύνομα ως προς την ανάθεση. Thank you. Well, that's exactly what I... Αυτό είπα ακριβώ. Δεν ήμασταν σε θέση να διαπιστώσουμε κάποια παραβίαση σε ό,τι φορά την ε, οδηγία 2004-17. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριο Γιά, τότε θα πρότεινα εγώ να κλείσουμε αυτή την αφορά και να το διαβάσουμε στον Ετούντα για ποιο λόγο και αντιστρόφως αν εκείνο επιθυμεί θεωρεί ή έχει επαρκείς ενδείξεις ή από λόγους να δώσει συνέχεια μπορεί να το πράξει ο ίδιος. Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε την αναφορά. Συμφωνώ με το ότι η αναφορά θα πρέπει να κλείσει, αλλά δύο σημείωσεις ε, να πω. Το ζήτημα των 25 ετών με ανησυχεί. Δεν νομίζω πως ε, ε, έχουμε συνάψει καμία συμφωνία 25 ετής διάρκειας με οποιαδήποτε επιχείρηση. Και το θέμα της αποτέφρωσης είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει ως πολιτική ομάδα. Να πω ότι μια που μιλάμε για τιμές και κόστος θα πρέπει να δούμε ποιο, ποιο είναι ο μέσος όρος ο κόστος ε, αναφερόμενος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η διαχείριση έχει ένα κόστος και αυτό το κόστος το πληρώνουν οι καταναλωτές. Αν υπάρχει λοιπόν μια κατάλληλη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, ένα παράδειγμα στην περιοχή που διαμένω ο πολίτης δεν επιβαρύνεται για, με το κόστος αυτής της αποτέφρωσης. Τώρα, σε ό,τι φορά την επιλεκτική ε, συλλογή των αποβλήτων και του σχετικού κόστους, να πω ότι θα πρέπει να δούμε ποια δυνατότητα υπάρχει για την διαχείριση των αποβλήτων Συμφωνώ πάντως με τον Στάλφο ότι αυτή η αναφορά θα πρέπει να κλείσει. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Το ζήτημα του κλεισίματος ε, πιστεύω θα βρει ανταπόκριση στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ε, υπογράμμισε ο συνάδελφος, ε, υπάρχει και το θέμα των ε, συμβατικών υποθέσεων όπως αυτή που συζητάμε χάρη στην αναφορά που υπέβαλε ο πολίτης αυτή η αναφορά για λόγω της μη αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών οργάνων και μη παραβίαση αυτή των ε, κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει να κλείσει λοιπόν η υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Προτείνουμε λοιπόν να κλείσει και να αποστείλουμε τα αίτια που μάθαμε σήμερα χάρη στη Συμβολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αναφερόμενο. Είχα ξεχάσει να πω στην αρχή ότι ο συναδελφό Μακμίλαν Σκότ θα ήθελε να συμμετάσχει στη συζήτηση για αυτή την αναφορά, αλλά είχε κάποιο πρόβλημα και δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται και ζητά συγγνώμη την απουσία του. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής ε, διάταξη 0768 του 2012 της Άννα Μαρίνα Βέλο, Ισπανικής Ιθαγένειας καταγγελία σε σχέση με εργασίες ε, χρυσορυχείου που πρόκειται να διεξαχθούν με τη μεδό της ανοιχτής εσκαφής στον Δήμο της Λακαμπάνα στη Γαλλικία. Δίνω λοιπόν το λόγο απευθείας στην αναφέρουσα για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Είμαι κάτοικος του Κορκοέστο, ενός χωριού της Γαλλικίας, που αυτή τη στιγμή ε, η επιχείρηση προβλέπει την εγκατάσταση ενός χρυσορυχείου ανοιχτού. Ε, αναφέρεται η προειδοποιώ ότι η τοποθεσία στην οποία θα εξεχνιαστείς απέχει μόλις 140 μέτρα από διάφορες τοποθεσίες της Natura 2000. Επίσης μιλάω για μια ιδιάζουσα περιοχή. Αυτό, αυτή η περιοχή πήρε τις απαραίτητες ε, άδειες ε, για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτή τη στιγμή όμως ε, δεν αναμένεται η κατάλληλη χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Θα αναφερθώ σε ένα πρόγραμμα, το αυτό το Edgewater, που στοχεύει στην καταστροφή 392 εκταρίων ατλαντικού δάσους στην Γαλλικία. Να πω επίση ότι η πλησφία των κατοίκων του χωριού και των γειτονικών χωριών Είμαστε κατά αυτού του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν ενωμένοι είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε το χρυσορυχείο να μην εγκατασταθεί εκεί. Καταρχήν είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με την γη. Πρόκειται για ένα περιοχή η οποία θα πρέπει να τύχει προστασίας για την επιβίωση των κατοίκων. Ε, πολλές ε, γενές γεννηθήκαμε ε, και μεγαλώσαμε με τα νερά του ποταμού αλλά και με το δάσος η γεωργία και η κτηνοτροφία επιτρέπουν στους κατοίκους την επιβίωσή τους. Έτσι έκαναν οι πατέρες μας, οι παππούδες μας και κάνουν το ίδιο τα αδέλφια μας και εμείς. Να πω ότι η κτηνοτροφία και η γεωργία παρέχουν τους απαραίτητους πόρους για την επιβίωση των πληθυσμών των χωριών. Τα ξενοδοχεία μας, τα οποία έχουν λάβει επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναπτύξει περαιτέρω την περιοχή. Οι επισκέπτες της περιοχής ε, αποτελούν το σημαντικό έσοδο για τις οικογένειες. Φτάνουν οι τουρίστες για να γευθούν τα τοπικά προϊόντα που βρώνονται από την θάλασσα και από την γη. Ο ορνηθολογικός τουρισμός κινηθεί. πολλοί έρχονται για να παρατηρήσουν ε, τα πτηνά τα οποία ζουν ε, στις εκβολές ε, του ποταμού. Επίσης επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή ξυλίας. Και να πούμε επίσης ότι τα δάση παρέχουν επίσης ε, και άλλα προϊόντα πέραν της ξυλίας. Το ορυχείο είναι ασυμβίβαστο με τις δραστηριότητες της περιοχής. Της περιοχής. οι εργασίες που προβλέπονται θα έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα επηρεάσουν τον, τον ποταμό Αγιόνσο. Η κατανάλωση 1,5 εκατομμυρίου κυβικών ε, μέτρων ύδατος θα καταστρέψει την ε, περιοχή. Όπως σας είπα, η τοποθεσία στην οποία θα εξευνούν απέχει μόνο 140 μέτρα από τις διάφορες τοποθεσίες Natura. μόνο ότι 230.000 υπογραφές έχουν κατατεθεί, δεν κατορθώσαμε να αλλάξουμε την άποψη των ε, υπευθύνων. Η πρόεδρος διακόπτη. Παρακαλείστε έστω και καθυστερημένα να μιλάτε πιο αργά και να ολοκληρώσετε. Ζητώ λοιπόν ε, μια δήλωση θεσμική λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό το πρόγραμμα στο Κορκουέστο. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η εκπρόσωπος της δεύτερης αναφοράς για το ίδιο θέμα. Ξέχασα να το πω προηγουμένως στην αρχή ότι είστε κι εσείς εδώ παρούσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το Φρανσίσκο Γαρτία Τρίγο για την εμπιστοσύνη και την πλατφόρμα για την προστασία του Κορκοέστο δε Δεμερκαντίνιος που μου ανέθεσαν να ε, παρουσιάσω αυτή την αναφορά. Σας έχει κάνει αναφορά μια έκθεση ε, με, ε, από πανεπιστήμιο του Σαντιάγου του Κομποστέλα που χαίρει μεγάλου κύρους για το αρσενικό που έχει βρεθεί στο Κορκοέστο. Δηλαδή το χρυσορυχείο, το έργο αυτό έχει υποτιμήσει ε, την διάχυση αρσενικού στη φύση και πόσο αυτό το χημικό στοιχείο που είναι άκρος ε, καρκινογόνο επηρεάζει την υγεία και το περιβάλλον. Το χρυσορυχείο όπως σας εξέθεσε ε, η αναφερόμενη θα έχει τεράστια καταστροφική και ολέθρια συνέπεια, θα καταστρέψει εκτάρια ολόκληρα όλα αυτά και στις δύο αναφορές ε, αναφέρονται εκτενώς ε, είναι δασικές εκτάσεις και ε, εκτατική γεωργία που πλήττονται αλληλεία, η δημόσια υγεία όλα αυτά ο Σάλο με υπογραφές πάνω από 250.000 κατοίκων 15-20.000 άνθρωποι διαδηλώνουν επανειλημμένα και έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος στη Γαλλικία τι σημαίνει αυτό το τεράστιο χρυσό ρηχείο ε, που ε, σχεδιάζεται. Είχα την ευκαιρία ως εκπρόσωπος του τοπικού κοινοβουλίου της Γαλλικίας το 12 και το 13 να αναφερθώ σε αυτό το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο στο Κορκόεστο, στη Ρος Μοντάνα, στη Χαλκιδική, στις Κουριές και ε, σε άλλα σημεία γονατίζουν μπροστά ε, σε καναδικές πολυεθνικές και άλλες ε, που έρχονται σε συγκεκριμένα μέρη για να διαφθείρουν, για να παρανομήσουν, για να ξεπεράσουν ε, τις ε, δηλώσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι copy-paste προηγουμένων αποφάσεων κυβερνήσεων, οι οποίες κυβερνήσεις υποκύπτουν σε αυτά τα συμφέροντα. Και γιατί τα λέω αυτά, δεν το λέει μόνο αναφερόμενος και εγώ εκπροσωπώντας τον, αλλά έχουμε δει και από την επιστημονική κοινότητα που τα έχει αναλύσει όλα αυτά, πώς η δήλωση περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων σχεδόν ταυτίζεται από ε, περίπτωση σε περίπτωση. Η εταιρεία ίδια κάνει τις ίδιες μελέτες παντού. Ε, ε, είναι η κοινωνική κατακραυγή. Ε, στα γαλλικιανά σας δείχνω εδώ το αυτοκόλλητο, λέω όχι στο χρυσορυχείο, στο κορκοέστο. Αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο πρόβλημα της Γαλλικίας, είναι πανευρωπαϊκό και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει και να υλοποιήσει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου του 2010 για την απαγόρευση ε, των, ε, και ανίων και άλλων ε, επικινδύνων ουσιών σε τέτοια έργα. Και πέρασε και στην έκθεση Χουντή μια δική μας τροπολογία την αναθεώρηση ε, για την οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ε, υπαίθρια ε, ορυχεία και αντίστοιχες εξωτερικές δραστηριότητες θα βγουν από το παράρτημα 2 και θα μπουν στο παράρτημα 1 ζητούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αν τηρηθεί η νομοθεσία το χρυσορυχείο στο Κορκοέστο δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για να διαχέεται αρσενικό στη φύση και να βλάψει την υγεία των πολιτών. Και μάλιστα κρύβονται πίσω από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αυτό είναι και κατά τη σύμβαση του όρχους και κατά τη ε, βούληση του τοπικού πληθυσμού. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βαλέιο Πέτραγκάλ. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε και στην ανακοίνωση της στη γραπτή του Μαρτίου 2013, ζήτησε πληροφόρηση για το θέμα αυτό, για τα χαρακτηριστικά του έργου και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίησή του, καθώς επίσης κατά πόσο συνάδει και σέβεται τις ε, ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα ζητήσαμε όλα αυτά από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει την απάντηση και κυρίως ε, συμπεριλαμβάνουν ε, κάποιες μελέτες του τοπικού Υπουργείου Περιβάλλοντος ε, της Περιφέρειας Γαλλικίας και άλλες αρχές Γαλλικίας. Λοιπόν, σύμφωνα με τις προφορίες αυτές, το έργο του Χρυσού του Κορκοέστο δεν έχει επιτραπεί, δεν έχει εγκριθεί και τώρα είναι σε διαδικασία για ε, επίλυση, σε άρνηση δηλαδή, απόρριψη του έργου. Και σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που μας διαβίβασαν οι Ισπανικές αρχές, σε περίπτωση που έρθει νέο αντίστοιχο έργο θα πρέπει και αυτό να ε, ε, υποβληθεί στην ισχύουσα διαδικασία και διοικητική και της αδειοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει καμία παραβίαση συνεπώς της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Σάνσες Πρισέντο. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τις δύο εκπροσώπους ε, των αναφερομένων Άννα Μαρτίνα Βαρέλα και Άννα Μιράντα. Πάντως νομίζω ότι είναι σωστό να απαντηθούν ε, οι αναφέρες. Ε, μπορώ να σας πω ότι δεν είμαι κάποιος που καταρχήν αντιτάσσεται στην λειτουργία ε, χρυσορχείων όπως συμβαίνει στην Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, ε, την Σουηδία. Οποιαδήποτε όμως δραστηριότητα εξόριξης θα πρέπει να σέβεται την κοινωνική νομοθεσία και να διασφαλίζει το οποιοδήποτε πρόγραμμα που κατατίθεται για στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γαλλικία που ε, επιδράζει μια περιοχή η οποία προστατεύεται από την Natura 2000 θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η υγεία των ε, πολιτών. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή έχει απαντήσει ότι περιμένει κάποιες απαντήσεις από τις εθνικές αρχές. Τώρα η Κομισιόν ε, έχει, μας έχει δώσει κάποιες προφορές που δεν περιέχονται στο φάκελο μας, ότι δηλαδή ε, προβλέπεται ήδη μια αρνητική απάντηση στην σχετική, για το σχετικό έργο. Νομίζω ότι το αίτημα των αναφερομένων καλύπτεται με την αρνητική αυτή εξέλιξη της ε, εγκατάστασης του χρυσορυχείου. Επίσης αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι κατά πόσον ένα έργο ε, είναι σύμφωνο με, με την κοινωνική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σχετικά προφορίες ε, και ως εκ τούτου αυτό το οποίο κρίνουμε είναι ότι το θέμα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό μέχρι ότου να υπάρξει μια απάντηση από τις ε, Ισπανικές αρχές όταν αν η απάντηση είναι αρνητική τότε ε, ε, θα είμαστε ικανοποιημένοι διαφορετικά θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κύριος Βιλμέγερ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις δύο κυρίες για τη δυνατότητα που έχουμε να μιλήσουμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών για αυτό το θέμα διότι όντως εγώ χωρίς να έχω ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούγοντάς σας σήμερα ερχόμουν εδώ να πω ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτό το πρόγραμμα, να ματαιωθεί. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Γαλλικίας θα δώσει αυτή την αρνητική απάντηση, ε, πράγμα που μας εξοικονομεί αρκετό χρόνο και πολύ περισσότερο την ε, ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική και κοινωνική βλάβη και ζημία. 322 εκτάρια δάσους, ε, φυσικός χώρος, ε, κτηνοτροφία, γεωργία, με το κιάνιο και το αρσενικό που χρησιμοποιείται στο χρυσορυγείο. Πραγματικά, από το Μάιο 2010 ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αντιταχθεί στη χρήση κιανίου για την εξόριξη χρυσού και σε υπαίθρια ορυχία. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Σάντσες Πρεσέδο παρά το γεγονός ότι δεν θα δοθεί η έγκριση όπως μας λέτε από τις αρμόδιες αρχές ε, ε, για καλό και για κακό όπως λένε στη Γαλλική ας την αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αφορά για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της για όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να ξέρουμε ότι τέτοια ορυχεία δεν θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, χαίρομαι για την απόφαση αυτή τη γαλλικιανής κυβέρνησης και ελπίζω να μην είναι συγκυριακή, αλλά είναι τέλεση ειδική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος. Ε, ε, ε Γκαρσία Γοήτια, τι πρόβλημα έχετε, εύκολο είναι το όνομά μου. ευχαριστώ. Συμφωνώ και με τον Ανατολή και με τον Βίλι Μέγε. Ε, για ε, τα όσα είπαν και για την κατάσταση και για το έργο. Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να έρχεται με οποιοδήποτε τίμημα και ιδιαίτερα όταν καταστρέφει την παραδοσιακή οικονομία και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής μιας περιοχής. Επιπλέον, για τις επόμενες γενναίες θα άφηνε μια πολύ επισφαλή κατάσταση για την οικονομική ανάπτυξη. Πέρα από το χρυσορυχείο αυτό το υπαίθριο που θα ήταν για κάποια χρόνια και μετά θα σταματούσε και θα άφηνε βλάβες ανεπανόρθωτες στο περιβάλλον. Επίζουμε η απόφαση των αρμοδίων αρχών της Γαλλικίας, δηλαδή η άρνηση της αδειοδότησης να ε, επιβεβαιωθεί. Ελπίζω να μην είναι παρελκυστική τακτική για να ξανάρθει το θέμα αυτό μετά από λίγα χρόνια. Πέντε χρόνια ισχύει η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να μην μας ξανάρθει μετά από μια πενταετία. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα θέματα αλλού. Διάφορα έργα που αναβάλλονται και επανέρχονται ανάλογα με την κοινωνική πίεση. Ευχαριστώ τις δύο αναφερόμενες και ε, ευχαριστώ και το λαό της Γαλλικίας για την κοινωνική πίεση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή αναφορών. Και αυτό είναι μια καλή απάντηση στον ευρωσκεπτικισμό. Μόλις ακούμε Ευρώπη να μην είναι αρνητικές οι σκέψεις που έρχονται. Παρακαλώ και εγώ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά μέχρι το θέμα αυτό να λυθεί οριστικά από τις αρχές της Γαλλικίας. Μέχρι να λάβουν την οριστική τους απόφαση λοιπόν εκεί και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή ε, μέχρι τη λήξη της δήλωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ κύριος ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις αναφερόμενες. Να πω καταρχήν ότι οι Ισπανικές αρχές όπως και η κυβέρνηση της Γαλλικίας ε, έχουν απόλυτη γνώση της ανάγκης ε, αποφυγής κάθε κινδύνου από τις εξορίξεις ε, ταυτόχρονα όμως ε, και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισπανίας, της Γαλλικίας προσφέρουν σε απαραίτητες ε, εγγύσεις τώρα. Σχετικά με τη συγκεκριμένη αναφορά και το είπε και ο πρόεδρος της περιοχής τον Οκτώβριο του 13 προ 3 μηνών ότι αυτό το σχέδιο δεν πρόκειται να ευοδοθεί. Σύμφωνα με τις προφορίες που έχω ήδη τον Ιούνιο 2013 αναφέρθηκε ότι το σχέδιο δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ούτε τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές κλπ. Έως εκ τούτου λοιπόν η, Γαλλή, η κυβέρνηση της Γαλλικής ε, ζήτησε απαραίτητες ε, εγγυήσεις, ε, υποχρεώσεις από πλευράς της επιχείρησης, αποδείξεις ότι θα τηρηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ανακοινώθηκε ήδη στην επιχείρηση η κατάργηση της, του έργου οι πληροφορίες που, που διαθέτω και είναι γνωστές και στα μέσα ενημέρωση της Γαλλικίας αλλά και στο τοπικό κοινοβούλιο και συμπίπτει με αυτά που μας ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το ε, έργο αυτό δεν πρόκειται να ευοδοθεί. Τώρα για τις ε, επιπτώσεις της περιβαλλοντικής το ζήτημα του κιανίου Ξέρω ότι το 93% των, των ε, προϊόντων που λαμβάνονται σε αυτά τα ορυχεία ε, δεν τη επεξεργασία με οικιάνιο, αν και πολλά ελέγχθηκαν. Να πω επίση κάτι ακόμα. Ότι η μελλοντική εγκατάσταση επεξεργασία δεν έχει πάρει τι απαραίτητε εγγυήσει, άδειε, συγγνώμη, αδειοδοτήσει και από πλευράς ε, αδειοδοτήσεων υπήρχαν εκκρεμότητες ήδη για λόγους περιβαλλοντικούς. Αναφέρομαι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ε, των, ε, των μετάλλων. Και επίσης είχε ζητηθεί μη ρήπανση των υδάτων κλπ και η σχετική επεξεργασία του φυσικά μετά από την χρήση. Έρευνα να υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δηλώσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτό το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση σύμφωνα με τους ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκή, την Ισπανική και την νομοθεσία της Γαλλικίας. Εντάξει, αν θέλετε να ε, περιμένουμε τις μερικές εξελίξεις, μπορεί να παραμείνει ανοιχτό το θέμα, αλλά ε, θα μπορούσε και να κλείσει εδώ. Ο κύριος Ζουργκάζη έχει το λόγο. Δεν θα πω πολλά. Ο κύριος Μιγιάν Μον τα ξεκαθάρισε, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Νομίζω δεν θα πρέπει τώρα να μπούμε σε στήρες συζητήσεις, Πρόεδρε, και να αναλωθούμε εκεί. Διότι όταν δεν υπάρχει έγκριση, όπως το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υφίσταται το θέμα. Αφού δεν του έχει δοθεί άδεια, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Και όπως είπε ο κύριος Μιγιάν, αν θέλετε να περιμένετε επίσημα να το ανακοινώσει η κυβέρνηση της Γαλλικίας, η τοπική, καλώς. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφέστατη, κατηγορηματικότατη για αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ο Πρόεδρος, οι κυρίες αναφερομένες έχουν το λόγο για να κλείσουν. Κυρία Μιράντα, ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Μέγε, εξ ε, και των δύο αναφορών και όλων των οργανώσεων και της πλατφόρμας που υποστηρίζει αυτό το θέμα της κατάργησης ε, της επένδυσης. Ευχαριστώ. Πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για διάφορους λόγους κατά την άποψή μας. Όχι μόνο με βάση τα επιχειρήματα ότι η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει πενταετή διάρκεια και στη συνέχεια μπορεί να επανέλθει το θέμα. Πολύ ωραίο το είπαν ορισμένοι βουλευτέ. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά δεν έχει υποθεί όλη η αλήθεια. Το έργο δεν εγκρίθηκε για λόγους οικονομικούς, διότι το ταμείο ήταν μείον, διότι έπεσε η τιμή του χρυσού και δεν ήταν ε, κερδοφόρο. Γιατί τη δήλωση ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν την είδαμε να αναγνωρίζει τους οικοτόπους των διαφορών ειδών που προστατεύονται. Παραλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς αυτό. Αυτό το λέγουν επιστήμονες ε, του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα, που είναι από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια ε, στην έρευνα, ε, στην εξόριξη. Εμείς δεν είμαστε κατά των ορυχείων, αλλά όχι τέτοιου είδους μεγαθύρια ορυχεία που ρηπαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε, η Επιτροπή σας το συζητάει και θέλουμε να ειδωθεί ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και υπάρχει ε, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2010 ε, που θα πρέπει να εφαρμοστεί για απαγορεύση του κιανίου. Τρεις μόνο ευρωπαϊκές χώρες το έχουν μεταφέρει στην νομοθεσία. Θα πρέπει να απαγορευτεί αυτή η ουσία γιατί υπάρχουν πολλές εκθέσεις για την επικινδυνότητά τους. Και, και όχι μόνο το κιάνιο και το αρσενικό. Και για το θέμα αυτό εγώ θα περιοριζόμουν από πλευράς του αναφερομένου της αναφοράς που εκπροσωπώ εγώ αλλά και της άλλης ε, θα έλεγα να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά μέχρι ε, ε, να λήξει η ισχύς της δήλωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή όχι τον άλλο μήνα όπως είπαμε αλλά την επόμενη πέντα αιτία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς το λόγο επ' αυτού. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όσα ακούσαμε από εσά, αποφασίζουμε λοιπόν να μείνει ανοιχτή, να παραμείνει η αναφορά για να δοθεί αυτή η συνέχεια όπως ακούσαμε στη συζήτηση και Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους αναφερομένους, τις αναφερόμενες ε, προκειμένου που μας ε, επέτρεψαν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ε, να μάθουμε και το νέο αυτό διαστόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι φρονεί αυτόν τον καιρό η κυβέρνηση της Γαλλικίας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι αναφορά υπαριθμών 10 στην ημερήσια διάταξή μας 0095 του 2012 του Χούλιο Μαρτίν Ντουχένο Μαγκλάνο και Χαβιέρ Καρίγιο Καστάνιο που εκπροσωπεί το κίνημα ΕΚΟ. Ποιοι είναι παρόντες εδώ αυτή τη στιγμή. Δύο είναι οι αναφορές ε, που έχουν συγχωνευτεί σε μία. Το ένα είναι από το Βαλτεμόρο Σπαρτάλ Εκολοχίστας σχετικά με τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βαλτεμόρο και Συμποσουέλος και το άλλο που εκπροσωπεί ο κ. Καρίγιο Καστάνιο για το ΕΚΟ είναι επεξεργασία λιμάτων και πάλι στη Μαδρίτη. Παρουσία λοιπόν των αφαιρωμένων θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καρίγιο για να μας εξηγήσει την αναφορά του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Αναφορών, ως εκπρόσωποι της κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης ΕΚΟ και Σπαρτάλ Βαλτεμόρο, που έχουν υποβάλει τις αναφορές θα θέλαμε και πάλι να διατρανώσουμε την πλήρη και κατηγορηματική μας απόρριψη και αντίθεση ε, στις μονάδες αυτές επεξεργασίας λιμάτων Μαδρίτε, Πούρα και Βαλτεμόρο. Πρόκειται για ένα σύνολο υποδομών που ε, θέλουν να τις εγκαταστήσουν σε προστατευόμενες ζώνες από διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκουν και στο δίκτυο 2000, Natura. Ε, χρειαζόταν περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Ε, υπάρχουν ε, προβλήματα στην πόλη του Βαλτεμόρα ως προς την επεξεργασία λιμάτων διπλασιάστηκε ο πληθυσμός περίπου την τελευταία δεκαετία και γι' αυτό χρειάζεται να γίνεται βιολογικός καθαρισμός από μια νέα μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Αλλά η πρόταση ε, της Μαδρίτης ε, ε, θέλουν να κάνουν είναι πολύ μακριά από το να λύσουν τα προβλήματα. Οπότε... Οι κατασκευαστές θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν εκεί τους σταθμούς, αλλά υπάρχουν προβλήματα δημόσιας υγείας ε, σύμφωνα με την οδηγία 92 43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα εδώ να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που αν περάσει ε, σημαίνει ότι θα καταστραφεί ένας βιότοπος που είναι ιδιαίτερης σημασίας και μοναδικός. Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα αντισταθμιστικά που από ό,τι φαίνεται ε, δεν έχουν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον νόμο σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι πάνω από 85% ε, του οικοπαίδου που έχει επιλεγεί ε, και από εκεί που θα περάσουν οι σωληνώσεις βρίσκονται σε οικοτόπους φυσικών, κοινοτικών ε, ενδιαφερόντων που ε, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακαιρεότητα του δικτύου Natura 2000 και μάλιστα ανεπανόρθωτες. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε όλους αυτούς τους οικοτόπους ε, αυτοί όλοι έχουν συμπεριληφθεί στον Εθνικό Μητρό του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ισπανίας για περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας έκουω και ε, η σε δράση που υπογράφουν αυτή την αναφορά λέμε ότι δεν έχει γίνει απαραίτητη ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ενώ στο πρόγραμμα του βιολογικού καθαρισμού στο Βαλτεμόρο δεν γίνεται σωστή διάγνωση στη μελέτη επιπτώσεων για το πώς ε, διακυβεύεται το περιβάλλον και η φύση. Επιπλέον σημαίνει αυτό ότι η μελέτη και η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του βιολογικού καθαρισμού έχει ξεπεράσει ε, τη διετία ε, που ισχύει και έχει λήξει. Και κανονικά σύμφωνα με την οδηγία θα πρέπει να γίνει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Εσπαρτάλ και το Ρόγια Τελακανάδα που βρίσκονται στο Βάλτε Μόρο και στο Σιέμπο Σουέλος φιλοξενούν ε, ε, ε, χλωρίδα και πανίδα ε, πολύ σημαντικών ειδών και συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000. Είναι στο κέντρο πραγματικά της Ιβερικής Χερσονήσου. Υπάρχουν διάφορα είδη φυτών, ενδυμικών που δεν απαντούν πουθενά άλλου στον πλανήτη, παρά μόνο εκεί. Και ε, ε, υπάρχουν ε, είδη που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον βότανολογικό, ζωολογικό και επιστημονικό. Θα θέλαμε τέλος να τονίσουμε την ύπαρξη εναλλακτικών τοποθεσιών για να κατασταθεί αυτός ο βιολογικός καθαρισμός. Κοντά στην προηγούμενη που περιορίζουν ε, την ε, περιβαλλοντική επίπτωση ενός έργου τέτοιας εμβέλειας και έχουν τεθεί υπόψη ε, της ισπανικής κυβέρνησης όταν είχε ανοίξει η διαβούλευση χωρίς να ληφθούν υπόψη. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, τώρα έχει έρθει η ώρα και ακόμα είναι γέρος να αναζητήσουμε μια λύση γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα έργα, δεν έχουν μπει θα πρέπει να ε, κλείσουμε λέγοντας ότι ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για το ενδιαφέρον τους, για το έργο τους και αν τελικά η εξέταση ε, των αναφορών μας δεν σας ε, δίνει αρκετά στοιχεία για να απορριφθεί αυτό το έργο ή οργανώσει που εμείς εκπροσωπούμε οικολόγηση δράση και έκου θα σας παρακαλούσαν, εάν το επιθυμείτε και το θεωρείτε σκόπιμο, να έρθετε να επισκεφτείτε τις εν λόγω περιοχές για να τα διαπιστώσετε αυτά οι δύο μας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ράμος Φλόριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ενώπιον δύο αναφορών του 2012 που συνδέονται με την επεξεργασία των ε, αποβλήτων στην ε, Ισπανία. Στην αναφορά 95 αναφερόμαστε στις αρνητικές επιπτώσεις ε, του προγράμματος Βαλτεμόρο στην Natura 2000 για το θέμα της αναφοράς 282 αφορά τους Δήμους Βαλτεμόρο και Συμποσουέλος και τον αρνητικό αντίκτυπο στο δίκτυο Natura 2000 για την παραβίαση οδηγίας και των οδηγιών εξοικοτόπους και τα Η άλλη οδηγία αναφέρεται στον δημιουργία υποδομών για την επεξεργασία λιμάτων στη Μαδρίτη. Επίσης ε, έχει ε, προωθηθεί από το κανάλι Ζαμπελ Σεκούντα το όταν έλαβε τις αναφορές η Ευρωπαϊκή η Κομισιόν αποφάσισε να κάνει μια έρευνα και απευθύνθηκε στις Ισπανικές Αρχές προκειμένου να λάβει τις παρατηρήσεις τους και τη θέση τους ε, για τα όσα κατάγελαν οι αναφερόμενοι και ε, ιδιαίτερα το ζήτημα της επίδρασης ε, το περιβάλλον. Αναφέρομαστε στην οδηγία 2011-92, η οδηγία η οποία κωδικοποιεί την οδηγία του άλλου 85 για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και με τις περαιτέρω τροποποιήσεις και την οδηγία για προσέγγιση τη φύση, ε, που οποία επανειλημμένα μας είχε απασχολήσει στην Επιτροπή, όπως η οδηγία για τα πτηνά και για τους οικοτόπους. Σύμφωνα με το άρθρο 6 οδηγίας για τους οικοτόπους χρειάζεται μια ε, κατάλληλη επεξεργασία. Τώρα για να, να πω ότι Υπάρχει και οδηγία 91 κάθετος 271 ε, για τα απόβλητα ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα μέτωπα ανοιχτά σε σχέση με την Ισπανία αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας ε, των ε, αποβλητών υδάτων. Το 2013 αυτό το θέμα ήταν αντικείμενο διάφορων ανταλλαγών επιστολών με την Ισπανικές Αρχές. Ε, η αρχική απάντηση όταν εξετάστηκε ε, αυτή, τη, ακολούθησε και ακολούθησαν άλλες ερωτήσεις για περαιτέρω διευκρινήσεις και θα πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με, την, με το Δήμο του Βαλτεμόρο έγινε οι περιβαλλοντικές, οι περιβαλλοντικές μελέτες και αυτή η διαδικασία ήταν υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτή η μελέτη επιπτώσεων οδήγησε στην μεταφορά της οδηγίας μια δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 8-2012 που διατέθηκε στο κοινό τον, το, ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν και οι Ισπανικές Αρχές διαπιστώσανε ότι σε αυτή την περιβαλλοντική μελέτη είχε δοθεί αντίγραφο των διαφόρων εκθέσεων που είχαν υποβληθεί. Έγινε επίσης ε, περιβαλλοντική μελέτη και να πούμε ότι το τμήμα αυτό της οδηγίας, ε, αυτής της ε, εκθέσεις για τα ύδατα Φυσικά αυτό δεν είναι και ένα λόγος ε, για να αποκλειστεί, ε, αποκλειστούν οι οδηγίες για έμπρουσες τη φύση. Παρατηρείται όμω ότι η οδηγία ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εφαρμογή των απαιτήσεων που προανεφέρθηκαν και που περιλαμβάνουν τι οδηγίε για την φύση. Υπάρχουν δυόμιση χιλιόμετρα σύνδεσης της ε, ΕΔΑΡ που είναι δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός. Οι Ισπανικές αρχές ε, χωρίσαν προφορίες σχετικά με τις μελέτες ε, που έγιναν αλλά και για τα διάφορα διορθωτικά μέτρα τα οποία ρίχθησαν επίσης μας εξήγησαν για τις ενδεχόμενες εναλλακτικές κάτι το οποίο μελετήθηκε κατά διάρκεια των μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων επίσης αποκλείστηκαν κάποιες ε, θέσεις ε, τοποθεσίες μάλλον για την εγκατάσταση αυτού του έργου. Επίσης εξετάσαμε τις προφορίες που μας έστειλαν οι αναφερόμενοι για τις επιπτώσεις σε κάποια ασπόνδυλα ζώα Νομίζω ότι αυτό δεν εμπίπτει στην οδηγία ε, ε, περί οικοτόπων, αλλά στην, σε άλλη οδηγία. Τώρα, σε όλη φορά το μόρο, οι τεχνικές υπηρεσίες της δεν ε, μπόρεσαν να διαπιστώσουν κάποια ε, παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Τώρα, για τα λίματα, 282, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε αναφορά συγγνώμη που αφορά ένα έργο Συρία που χρησιμοποιεί το λιμάνι των δύο Βαλτεμόρων στην αυτόνομη περιφέρεια τη Μαδρίτη. Η Επιτροπή λαμβάνει των Ισπανικών Αρχών και ειδικότερα τι εκθέσει που εκπώνησαν η κυβέρνηση τη αυτόνομη περιφέρεια τη Μαδρίτη, καθώ επίση και η δημόσια επιχείρηση Κανάλ Ντεζαμπέλ 2, η οποία αποτελεί και τον φορέα υλοποίηση των λόγω έργων διαχείριση των λιμάτων. Οι Ισπανικές αρχές ε, απαντώντας ε, στο αίτημα ε, περαιτέρω πληροφοριών της ε, της Κομισιόν ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα περιόριζαν σημαντικά τις επιπτώσεις στο την, την οδηγία Natura 2000 ε, τώρα. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές η επαναχρησιμοποίηση των αστικών κλιμάτων θα ξεκινούσε το τέλη 2013 αλλά τα έργα δεν έχουν, σχετικά έργα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τώρα για να συμπλούσω την πληροφόρηση δεν προβλέπεται κοινωνική χρηματοδότηση για κανένα από αυτά τα προγράμματα, ούτε επίση προβλέπεται κάποια χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα, για να ολοκληρώσω την ενημέρωση, οι υπηρεσίε Κομισιόν δεν μπόρεσαν να ε, διαπιστώσουν ότι υπήρξε παραβίαση του κοινωτικού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Ιρασάβαλ Μπέιτια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφερομένους που ήρθαν εδώ να μας πούν για το θέμα αυτό. Έχω μια ερώτηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασικά, γιατί αν κατάλαβα καλά, κάποιον από τους αναφερομένους είπε ότι η μελέτη, η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει λήξει. Από πλευράς κοινοτικού δικαίου αυτό έχει επιπτώσεις ε, σε αυτό που μόλις μας είπατε, ερώτηση. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου και τη νομική δηλαδή, αυτό δεν έχει επίπτωση. Δεν ε, υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια των δηλώσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των ε, αναφορών των εκθέσεων όπως αναφέρεται στην οδηγία ή του ψηφίσματος. Αυτό το όριο το θέτουν ε, ορισμένες κρατικές νομοθεσίες. Ε, όπως στην Ισπανία ας πούμε, ακόμα και κάποιες περιφερειακές νομοθεσίες των αυτονόμων περιφερειών δεν, για την οδηγία δεν υπάρχει χρονική διάρκεια. Μπορεί να είναι επιπλέον στοιχείο ή επιχείρημα για να ε, ζητηθεί από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές να δοθεί απάντηση. Και το κάνουμε γιατί όταν αργούν πολλοί να δώσουν την περιβαλλοντική τους μελέτη ρωτούμε αν υπάρχουν νέα δεδομένα, ε, αλλαγή του δικτύου 2000 κτλ. Ευχαριστώ και άλλη ερώτηση ο κύριος ε, η Ρασαβαλμπέιτια για τη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων και αυτό που προτείνετε εσείς ως εναλλακτική λύση είπατε ότι το έχετε μελετήσει αυτό που προτείνουν και έχει απορριφθεί διότι αυτό θα σήμαινε μεγαλύτερο κόστος λόγω άντληση των υδάτων. Αυτό είναι αμυγό οικονομικό επιχείρημα μπορείτε να το αντικρούσετε με διαφορετικό τρόπο. Έχετε και άλλη ερώτηση, λέει ο κύριος Μέγερ, για να τη σωματοποιούμε λίγο. Ε, όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ε, οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποχρεώνει τα κράτη-μέλη και οι αντίστοιχε οδηγίε για τη φύση είναι να μελετούν διάφορα εναλλακτικά ε, προγράμματα ε, διότι η αρχική πρόταση όχι η νέα που αναθεωρείται τώρα ε, η αρχική είναι ότι αν έχει μελετήσει διάφορες εναλλακτικέ λύσεις στο κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώσει ε, για τα διάφορα αυτά εναλλακτικά σχέδια και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις ε, για το περιβάλλον από τα διάφορα έργα. Βεβαίως το ε, οικονομικό επιχείρημα από μόνο του δεν ισχύει δεν ευσταθεί. Αλλά αν καταλήξουν οι αρμόδιες αρχές ότι η εναλλακτική λύση που επελέγει δεν έχει σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που έχουν τα κράτη-μέλη όταν λαμβάνουν ε, αποφάσεις. Τώρα άλλο θέμα θα ήταν να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις και να ε, φαίνεται σαφώς ότι η μία βλάπτει το περιβάλλον και να επιλεγεί αυτή μόνο για οικονομικούς λόγους και κόστους και τίποτα άλλο. Αλλά τα κράτη-μέλη με την οδηγία αυτή για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν μια στοιχειώδη δυνατότητα, περιθώριο λιγμών για να αξιολογούν την κατάσταση. Α, θέλετε να συνεχίσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής Γι' αυτό ζητώ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Εάν το οικονομικό κόστος της εναλλακτική λύσης που προτείνουν οι αναφερόμενοι που δεν, έχει καμιά περιβαλλοντική επίπτωση είναι πια τόσο μεγάλο ε, απέναντι στην εναλλακτική λύση που προτείνουν οι Ισπανικές αρχές. Τόσο μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές τα οικονομικά επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ακριβώς ε, εις βάρος του περιβάλλοντος και με τρόπο πολύ ελαστικό, σαν μαστίχα είναι ελάστιχο. Και για να στραφούν ή να διοχετευτούν ε, τα αποτελέσματα προς μια συγκεκριμένη κατάσταση για να ευνοηθούν ορισμένοι. Γι' αυτό ρωτάω. Ε, τελευταίος έχει το λόγο ο κύριος Καριό Καστάνιο που υπέβαλε την αναφορά. Mm. Αν δεν σας πειράζει να απαντήσω εγώ, είμαι μέλος ε, των οικολόγων σε δράση του Βαλντεμόρο, που είναι η άλλη οργάνωση. Ακούστε και ότι η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων θα έχει επιπτώσεις, οι σωλήνες δηλαδή, το δίκτυο, σε ε, μια περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και ισχυρίζονται ότι δεν πειράζουν το βιότοπο. Δεν ισχύει καθόλου. Είναι ε, οικότοποι προτεραιότητας, ενδυμικά είδη, πάρα πολύ πολύτιμα ε, και είναι υφάλμηρα τα ύδατα. Τα έχουμε όλα αυτά ε, τεκμηριώσει και αν δεν αρκούσε αυτό υπάρχουν και τα πρακτικά των δασικών αρχών της κοινότητα κοινότητας Μαδρίτης, περιφέρειας. Άλλο θέμα που αναφέρθηκε ήταν πόσο ισχύει η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όντως, σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία και την τοπική της ε, περιφέρειας Μαδρίτης, προβλέπεται όταν έχει λήξει η μελέτη αυτή να γίνει νέα ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εμείς έχουμε φέρει τεκμηρίωση η οποία στοιχειοθετεί ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει διεξαχθεί με το σωστό τρόπο. Και ήρθαμε και αποδείξαμε ότι ε, είναι πραγματικά ε, υψής του οικολογικού ενδιαφέροντος ε, οι περιφέρειες που θα κατασταθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα για το πού θα εγκατασταθεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού ή επεξεργασίας λιμάτων, ε, ε, αυτό που προτείνουμε εμείς έχει πολύ μικρή διαφορά. Και αν χρειάζεται σταθμός άντλησης υδάτων, σε σχέση με την άλλη μελέτη που δεν το προβλέπει, άλλαξε το έργο και έχει συμπεριλάβει πλέον ε, μονάδα άντλησης ε, ακριβώς ε, εκεί σε ευαίσθητες οικολογικές περιοχές χωρίς την αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ πολύ. εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, θα μιλήσω όχι ως πρόεδρος, αλλά ως βουλευτής της Ενωτικής Αριστεράς από την Ισπανία, να σας πω την άποψή μου και μετά να κάνω μια πρόταση. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Ιρασάμπαλ Μπέιτια, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Όντως, η συζήτηση που μας απασχολεί έχει ως εξή. Σε κοινωνικό επίπεδο κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνει μια μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Το θέμα είναι πού θα κατασκευαστεί έτσι. Να μελετήσουμε λοιπόν τα εναλλακτικά δεδομένα που έχουν, το κόστος που έχουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι βιώσιμη αυτή η μονάδα, να λαμβάνει υπόψη την περιοχή και τη ζώνη ε, που πρέπει να διαφυλαχθεί στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Αυτό το θέμα γίνεται και στην τοπική βουλή της Μαδρίτης και η δική μου πολιτική ομάδα εκεί έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες που ακόμα είναι ανοιχτές και κοινοβουλευτικές και κοινωνικές. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να δούμε, να μελετήσουμε την εναλλακτική λύση. Αυτά. Και τώρα μιλώ ως πρόεδρος και θέλω να πω ότι με βάση τα όσα ακούσαμε και όπως διεξήχθη η συζήτηση, συμφωνώ με τον κύριο Ιρασά Μπαλμπέιτια που ζητάει να παραμείνει ανοιχτό το θέμα και να έχουμε και νέα πληροφόρηση για να καταλάβουμε τι γίνεται με τις εναλλακτικέ λύσεις. Να παραμείνει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά και να γίνει αυτή η παρακολούθηση για τα εναλλακτικά έργα. Συμφωνούμε. Για να πέρασουμε στην επόμενη αναφορά και ευχαριστούμε τους αναφερομένους και τους ε, προσώπους της ΕΚΟ και των οικολόγων εν που μας φέρανε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Αναφορών. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αναφορά υπαριθμών 11. Παρίσταται ο αναφερόμενο. Είναι η αναφορά του κυρίου Βασίλη Χατζη Ευαγγέλου Κυπριακής Ιθαγένειας σχετικά με εικαζόμενε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Απουσιάζουν οι αναφερόμενοι, οπότε θα δώσω μέσα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με το προφανές ζήτημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να παρεμβούν μόνο σε ζητήματα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα δύναμη των συνθήκων και ιδιαίτερα σύμφωνα με το, το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμοζεται μόνο στο πλαίσιο της ενωτικής νομοθεσίας ε, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη μελετήσαμε και ξαναμελετήσαμε το ζήτημα Στείλαμε δύο απαντήσεις, ε, συμβουλευτήκαμε διάφορες ε, υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τα στοιχεία που συλλέξαμε δεν μπορούμε να βρούμε τη σύνδεση μεταξύ του ζητήματος που υποβάλλει ο αναφερόμενος και το δίκαιο. Μας φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα αφορά το δικαίωμα ιδιοκτησία να υπενθυμίσω ότι το άρθρα 3, 4 και 5 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας αποτελεί θέμα εθνικής αρμοδιότητας με την επιφύλαξη των εθνικών ε, διατάξεων για το δικαίωμα ιδιοκτησίας από τα στοιχεία που συλλέξαμε, η προκειμένη υπόθεση είναι καθαρά εθνικής αρμοδιότητας. Φυσικά κάποια ζητήματα που απορρέουν από το δικαίωμα ιδιοκτησίας μπορεί να έχουν στοιχεία ώστε να εμπίπτουν ε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά αυτή η σχέση πρέπει να αποδειχθεί. Ε, κατά πόσο υπάρχουν, για παράδειγμα, διασυνοριακά χαρακτηριστικά ή κατά πόσο ε, υπάρχει περίπτωση παραβίασης διατάξεων ή νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπερασματικά λοιπόν εμείς δεν βρήκαμε τέτοιο, δεν εντοπίσαμε τέτοια σύνδεση μεταξύ του ζητήματος αυτού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Συνεπώς δεν μπορεί να συνεχιστεί ε, άλλο η αναφορά αυτή Υπενθυμίζουμε ότι αν ο αναφερόμενος ε, θεωρεί ότι τα δικαιώματα του παραβιάζονται, φυσικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί μια δυνατότητα προσφυγής ε, αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα ε, τοπικά χώρια ένδικα μέσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανεί το λόγο από του συναδέλφους ε, βουλευτές. Θεωρώ λοιπόν ότι... Μάλλον το πω Ξέρουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε παρακολουθήσει το θέμα και η Επιτροπή μας για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι το θέμα είναι αρκετά ευαίσθητο ώστε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η ε, αναφορά, δηλαδή να παραμείνει ζητώ για να βάλουμε περισσότερες προφορίες και να δώσουμε τη συνέχεια που αρμόζει. Ευχαριστώ πολύ. Περνούμε στην τελευταία λοιπόν αναφορά. 1653 το 2010 της κυρίας Μαρκέλα Ισαΐα Τσιάκα, Κυπριακής Ιθαγένειας, εξ ονόματος Κυπριακής Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μητέρων, σύμφωνα σχετικά με διακρίση βάρος παιδιών, γυναικών και προσφύγων. Δεν έχουμε εκπρόσωπο εδώ των, της αναφερομένης. Ε, θα πάρει το λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ηλιόπουλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην καταπολέμηση κάθε μορφή διακριτική μεταχείριση ε, δύναμη των εξουσιών που τις χορηγούνται από τις συνθήκες, τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη αξία ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Ωστόσο, ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων εφαρμοστεί στα κρατη μόνο κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ισότητα των Φύλων καλύπτει την κοινωνική ασφάλιση, την απασχόληση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε. Αυτού του τρει τομεί. Όσον αφορά λοιπόν την παρούσα αναφορά, Είχαμε εκτενή αλληλογραφία με την αναφέρουσα, η οποία υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Κομισιόν, την οποία κλείσαμε. Για ποιο λόγο θα εξηγήσω τώρα. Όπως φαίνεται, η διαφορετική μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην παρούσα υπόθεση καλύπτει κοινωνικά ε, κοινωνικές παροχές που δεν αποτελεί αντικείμενο της ε, οδηγίας για ε, την ισότητα των φύλων. Κοινωνικά επιδόματα λοιπόν αυτά δεν καλύπτονται από το ενωσιακό δίκαιο. Τα κρατημέλη είναι εκείνα που πρέπει να τηρούν τι υποχρεώσει του για τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω αυτά απορρέουν από το διεθνέ δίκαιο. Γι' αυτό τον λόγο παραπέμψαμε την αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ζήτησε τον λόγο, παρακαλώ. Όπως καταλαβαίνω αυτό δεν εντάσσεται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων, τας, αρμοδιοτήτων μας, αλλά μπορούμε να αφήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή όσο του λάβουμε απάντηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έχουμε απομείνει από βουλευτέ εδώ ο κύριο Βαλένσα και εγώ, οι εξή δύο. Ε, δέχομαι και εγώ την πρόταση του κυρίου Βαλένσα υπό την έννοια και ισχύει και το ίδιο ε, που είπα στην προηγούμενη αναφορά, είναι αρκετά ευαίσθητα τα θέματα αυτά, ώστε να ε, είμαστε σε θέση να ζητήσουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να παρακολουθήσουμε την πορεία της. Μου λέγουν από τη Γραμματεία ότι μπορούμε να διαβιβάσουμε και στην Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα αυτό για να το παρακολουθούν και εκείνοι παραλλήλως. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό το θέμα ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση της Επιτροπής μας μέχρι τις 5.30 όπου ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ όλους σας και τους διερμηνείς ε, και τις διερμηνείς καθώς και τους αναφέροντες.